Der Präsident! Uiuiui, mein lieber Mann. Guten Tag, meine Damen und Herren. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ.